Buenas tardes. Καλό σας απόγευμα. Συνεχίζουμε λοιπόν την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής Αλίας. Έχουμε το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη που είναι η παρουσίαση από το θεματικό τμήμα Β μιας μελέτης για την συμβατότητα των εισαγωγών προϊόντων αλίας όσον αφορά και την υδατοκαλλιέργεια με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κονσόρσιο Γκόπα είχε δοθεί αυτή η γνωμοδότηση και οι ερευνητές και σε σχέση με τη σύνταξη της μελέτης έχει διανεμηθεί ήδη αυτή η μελέτη σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Αλίας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι άμεσα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλωσορίσουμε τους εισηγητές ε, <clears throat> τον κύριο Κάρλος Πέιλιν και την κυρία Σαλίν Γκοντάν, εκπροσώπων της ομάδας πολιτικών συμβούλων Κονσόρσιο Κόπα Γκόπα και που θα μας ενημερώσουν για αυτή τη μελέτη. Ο κύριος Πάλιν έχει πρώτος τον λόγο. Παρακαλώ. thank you very much. Um, good afternoon, everyone. My name is Carlos I'm presenting this. Καλησπέρα σας. Παρουσιάζω την ε, μελέτη που μόλις ε, είπε ο Πρόεδρος ε, ότι θα σας παρουσιάσω. Είναι η Σαρλίν Κοντά μαζί μου, η οποία συμμετείχε και εκείνη στις εργασίες. Οι άλλοι δύο σύμβουλοι που συμμετείχαν δεν είναι εδώ σήμερα. Θα κάνω μία σύντομη παρουσίαση ε, για τα πορίσματα της μελέτης αυτής ε, θα είδατε ότι υπάρχουν και συστάσεις που έχουμε συμπεριλάβει στην έκθεσή μας. Ε, δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες για τις συστάσεις αυτές στην παρουσίασή μου, γιατί τα πορίσματά μας οδηγούν καταλογικό τρόπο σε πολλές συστάσεις. Υποθέτω ότι είχατε το προνόμιο να διαβάσετε την έκθεση ήδη, οπότε δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες. η εμβέλεια της ε, έκθεσης ε, ήταν να αναλύσουμε ε, την διαδικασία των εισαγωγών των προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας βάσει υγειονομικών μέτρων και σε σχέση με την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία. Μας συζητήθηκε να διερευνήσουμε το βαθμό στον οποίο τα αλλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας είναι συμβατά με την Ευρωπαϊκή ε, Υγειονομική Νομοθεσία. Επίσης έπρεπε να εντοπίσουμε κάποια σοβαρά ζητήματα και να προτείνουμε συστάσεις. Πρόκειται λοιπόν για μια μελέτη η οποία σκοπό έχει να τροφοδοτήσει τη συζήτηση ε, για τα ε, θέματα που μας ζητήθηκε να καλύψουμε. Δεν είναι μία μελέτη η οποία σκοπό έχει να αναθεωρήσει την ομοθεσία ε, στις λεπτομέρειές της μπορεί να υπάρξουν ε, κάποιες συνέσπιες ως προς αυτή την κατεύθυνση αν η Επιτροπή σας και άλλες επιτροπές ε, το θεωρήσουν αναγκαίο αλλά εμείς δεν θα μπούμε στην ουσία της νομοθεσίας για να πούμε κατά πόσο θα πρέπει να διατυπωθεί καλύτερα ή ακριβέστερα το ένα ή το άλλο τμήμα της νομοθεσίας. Η μέθοδος ε, που ακολουθήσαμε ήταν αρκετά ασυνήθις. Χρησιμοποιήσαμε στατιστικά από την Eurostat και από άλλες πηγές για να δώσουμε την εικόνα των διεθνών αγορών αλλιευτικών προϊόντων. Είχαμε και κάποιες δευτερεύουσες ε, πηγές, ε, δηλαδή ερωτηματολόγια που στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στις υπηρεσίες τους ε, στα κράτη-μέλη. Ε, ήρθαμε σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, ε, με το, την Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων στην Ιρλανδία, με την Υπηρεσία Ελέγχου των Τροφίμων και πολλούς άλλους φορείς. Προσπαθήσαμε λοιπόν να, δήσουμε να δούμε κατά πόσο υπάρχει συμβατότητα με τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν τα προϊόντα αυτά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν είναι συμβατά με τα μέτρα. Ε, μελετήσαμε κυρίως τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Ε, Χρησιμοποίησαμε την εμπειρία μας σε σχέση με τρίτες χώρες που εξάγουν προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης σε 79 χώρες ε, ΑΚΕ ε, και ΟΣΑ. Είδαμε δηλαδή ε, ποια, ποιες εισαγωγές υπάρχουν βάσει των προγραμμάτων που έχουμε με τις χώρες αυτές και 50 προγράμματα τα οποία καλύπτονται και πάλι από την ΤΕΒΚΟ σε σχέση με την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας για την παράνομη λαθρεία και άναρχη αλία ε, στις τρίτες χώρες. Τα διεθνή ε, προϊόντα, τα διεθνή αλληλευτικά προϊόντα το διεθνές εμπόριο συγγνώμη, στα αλληλευτικά ε, προϊόντα είναι Επίσης είναι πολύ σημαντικό ε, σε σχέση με τον καφέ, το κακάο, την, ε, το, ρύζι, το κρέας, ε, τις μπανάνες, τη ζάχαρη. Βλέπετε ότι τα αλλιευτικά προϊόντα είναι, έχουν μεγαλύτερο όγκο από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που σας ανέφερα. Επίσης θα δείτε ότι η ποσότητα, η αξία του εμπορίου έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό σας το λέω για να τονίσω τη σημασία του εμπορίου ε, στα ε, αλλιευτικά προϊόντα. Από ε, πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπετε σε αυτό το γραφικό, σε αυτή τη γραφική αναπαράσταση, ότι η αυτάρκεια έχει μειωθεί πολύ. θα μπορούσα να βάλω 40 με 60 τότε θα ήταν ε, πολύ μεγαλύτερη η μείωση που θα βλέπατε, γιατί ουσιαστικά η αυτάρκεια έχει μειωθεί από 60% σε 40% η αυτάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα προϊόντα λίας και υδατοκαλλιέργειας. Έχουμε δηλαδή μια αυξανόμενη εξάρτηση ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενα προϊόντα. Η φύση των προϊόντων αυτών και ο προορισμός τους ε, ε, ποικίλει. Ε, βλέπετε ότι η Ισπανία ε, είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας, μετά η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και ούτω καθεξής. Όλοι οι υπόλοιποι, όλες οι υπόλοιπες χώρες μετά την Πολωνία είναι απλώς ένα κλάσμα αυτού που μόνη της η Ισπανία εισάγει. Οπότε λοιπόν ε, οι εισαγωγέ ε, αφορούν κυρίω κάποιε συγκεκριμένε χώρε που τι ευνοούν και βλέπετε επίση ότι η φύση των εισαγωγών, δηλαδή βάσει του τελωνιακού κώδικα, μόνο αυτά τα χρώματα μπορείτε να, να, να δείτε για να καταλάβετε ε, πόσο επικοινόμορφη είναι αυτή η αγορά. Από πού προέρχονται τώρα οι εισαγωγέ αυτές, από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι που προερχονται τωρα οι εισαγωγε αυτες απο τριτες χωρες εκτος ευρωπαικης ενωσης και αυτο ειναι προσπαθουμε να εξετάσουμε στη μελέτη, Νορβηγία, Κίνα, Βιετνάμ, Ηνωμένε Πολιτείε κυρίω. Όμως θα δείτε επίσης ε, ότι η προέλευση των προϊόντων είναι πολύ πιο, παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία από τον προορισμό. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, η στήλη λυπή είναι πάρα πολύ ε, σημαντική. Τώρα, το τι εξάγουν οι διάφορες χώρες επίσης παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλία. Να περάσω τώρα στη, στα πορίσματα που αφορούν ε, την, ε, ε, τα υγειονομικά και την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων αυτών. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε όλοι ότι το πακέτο για την υγεία είναι ένα πακέτο το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κανονισμός ε, για την παράνομη λαθρέα και αλλαρχιαλία είναι πρόσφατος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβει κάποιος υπόψη όταν βλέπει τις παρατηρήσεις ε, και τα πορίσματα της έκθεσης. Ε, το ένα από τα δύο είναι σχετικά όριμο και το άλλο είναι μάλλον ε, πρόσφατο και συνεπώς ε, δεν έχει εξελίξει τις διαδικασίες του ακόμα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι από πλευράς υγιεινής η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα ε, σωστό πλαίσιο για τις χώρες, τις τρίτες που θέλουν να ε, κάνουν εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η λογιστική έλεγχη του FVO, του Γραφείου Κτηνιατρικών Θεμάτων και Τροφίμων, είναι αυστηρό και κάνει καλούς ελέγχους σε σχέση με τα προϊόντα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε την κατάσταση στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ιαπωνία και είδαμε ότι και στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία επικοινωνία έχουν ε, συστήματα ανάλυσης του κινδύνου για να εξασφαλίσουν ε, την, ε, την καλή ποιότητα εισαγωγή αλλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Υπάρχουν λοιπόν εγγυήσει από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο τη νομοθεσία ότι αυτά τα προϊόντα που εισάγονται σε αγορέ Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφώνονται με τι προδιαγραφέ υγιεινή. Σύγκριση τώρα των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτων μελών και των δυναμικών του συστημάτων δείχνουν παρόμοιες ε, προδιαγραφές που ισχύουν ε, και στις δύο ομάδες. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί η υγιεινή και ε, η ποιότητα ε, βάση της νομοθεσίας σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν ε, ίσες προδιαγραφές ε, στις χώρες που θέλουν να κάνουν εξαγωγές σε ευρωπαϊκές αγορές, όπως επίσης και με την νομοθεσία που οι ίδιες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εφαρμόζουν. Τα κράτη-μέλη όμως και οι έλεγχοι τους ε, δεν είναι εναρμονισμένα πλήρως ε, ε, και μιλάω κυρίως για τον έλεγχο μέσω των πιστοποιητικών υγείας, προϊόντα, προϊόντα σκαφών με ευρωπαϊκή σημαία δεν, έχουν πάντοτε, δεν την χάνουν πάντοτε των ιδίων ελέγχων με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα. Ε, υπάρχουν διαφορές, ε, για παράδειγμα, στη θεώρηση από τα κράτη-μέλη του τι θα πει ένα, στόχο, ένα ε, μακρινών αποστάσεων. Και αυτό έχει βέβαια αποτέλεσμα ε, ως προς τα αλλιεύματα που υπάρχουν σε ένα σκάφος ε, με μια συγκεκριμένη σημαία. Επομένως, ο στόλος μακρινής απόστασης, ε, που είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τα αλλιεύματα, με τα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και συνεπώς δεν υπόκειται στους, ολόχους στους ελέγχους, στα σημεία ε, ε, ελέγχου τα μεθοριακά, που είναι κάτι το οποίο ισχύει για εισαγωγές από τρίτες χώρες. Ε, τα συστήματα ελέγχου των τροφίμων επίσης είναι, συμμορφώνονται σωστά με, την νομοθεσία. Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά ε, την έλλειψη των ε, σωστών αρμόδιων αρχών ε, με αρκετά κατηρτισμένο προσωπικό σε σχέση με την λειτουργία των εργαστηρίων και σε μερικές περιπτώσεις σε σχέση με την ανιχνευσιμότητα πρώτων υλών. Υπάρχουν λοιπόν ακόμη κάποια προβλήματα ε, όμως ε, εφαρμόζονται ε, πολλά μέτρα. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν προγράμματα δωρητών, προγράμματα εκπαίδευσης, τεχνική υποστήριξη και επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα σε μια προσπάθεια συμμόρφωσης με το πακέτο για την υγιεινή. Υπάρχει επίσης ένα σύστημα ε, έγκαιρης προειδοποίησης για το πακέτο αυτό και δείχνει ότι δεν απειλείται η υγεία των καταναλωτών από τα ε, προϊόντα αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Το σύστημα αυτό είναι ε, αποτελεσματικό, αλλά η χρήση του δεν είναι πάντοτε συστηματική από τα κράτη-μέλη οι αποφάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τον περιορισμό εισαγωγών ε, από κάποια συγκεκριμένη χώρα βάσει κάποιας ανάλυσης που κάνουν για τον κίνδυνο από τη χώρα αυτή λόγω κάποιων στοιχείων που μπορεί να βρέθηκαν στις εισαγωγές μερικές φορές είναι αυθαίρετοι και όταν οι έλεγχοι στα F, ε, του FVO στα κράτη-μέλη και στις τρίτες χώρες έχουν εντοπίσει προβλήματα, πολλές φορές ε, η παρακολούθηση ε, είναι κάπως κατακαιρματισμένη. Για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν η σύνοψη των πορισμάτων μας για το θέμα το υγειονομικό. Όσον αφορά τώρα την παράνομη αλληλεία, να συνεχίσω με τη μελέτη μας, ε, η παράνομη, λαθρέα και άναρχη αλία παίρνει διάφορες μορφές. Ε, βλέπετε μια γραφική παράσταση των διαφόρων μορφών που μπορεί να λάβει, αλλά βλέπετε είναι μόνο δύο διαστάσεων αυτή η προσέγγιση για κάθε περίπτωση παράνομης ή ε, ε, λαθρέας αλίας ε, υπάρχουν διάφορα είδη εξοπλισμού που μπορεί να απαγορεύονται, υπάρχουν περιορισμοί περιορισμοί για την περίοδο, ως προς την περίοδο αλίευσης για παράδειγμα και πολλοί άλλοι τρόποι. Ξέρω ότι τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα στην Επιτροπή. Ε, λέω ότι γίνεται υποτίμηση των ε, ε, αλλιευτικών πόρων και ότι αυτό βέβαια έχει βεβαίως μεγάλο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Οι εισαγωγές πάρα πολύ επηρεάζονται από την παράνομη λαθρέα άναρχη αλία. Ένα εκατομμύριο ένα δισεκατομμύριο ε, σε έσοδα χάνονται ε, κάθε χρόνο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ευάλωτη και σε, εσωτερικέ και σε, και σε εσωτερικές και εξωτερικές περιπτώσεις παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει πόσο σημαντικό είναι το πιστοποιητικό αλλιεύματος το οποίο υπογράφουν τρίτες χώρες και επιστοποιεί ότι προέρχονται από νόμιμη πηγή αυτά τα αλλιεύματα. Δεν θα σας πω τίποτε καινούριο αν σας πω ε, ότι κάποια κράτη-μέλη ε, ε, έχουν ε, είναι, είναι αντικείμενο ελέγχων ε, και, από, ε, και διεθνών και εθνικών. Μερικά κράτη-μέλη έχουν κακές επιδόσεις στον τομέα αυτό και μερικές φορές συμμετέχουν σε παράνομη λαθρέα και αναρχιαλία και αυτό το βλέπουμε και στον τύπο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στο πλαίσιο της δικής μας ε, μελέτης, εκτός των κοινοτικών υδάτων, ε, όταν ε, οι, δεν μπορούν να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του κράτους, των ελέγχων του κράτους σημαία ή του παράκτιου κράτους ή του λιμένα. Όσον αφορά τον κανονισμό τώρα για την ε, παράνομη λαθρέα και άλλη αρχαιαλία, είναι πάρα πολύ σωστό το πλαίσιο του, αλλά υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή του. Ε, μερικές, ε, μερικά τμήματά του είναι κακώς διατυπωμένα και σε μερικές περιπτώσεις ε, ε, ερμηνεύονται οι διατάξεις από ε, τρίτες χώρες με διαφορετικό τρόπο από ό,τι χώρες εισαγωγής και συνεπώς κάποια φορτία μπορεί να χάνονται με αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες εσόδων λόγω διαφορές στην ερμηνεία του κανονισμού αυτού. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ε, επικρίνουν ε, κάποιες πτυχές του συστήματος. Φαίνεται να υπάρχουν όμως ε, λίγες αποδείξεις σε επίπεδο κοινοτικό. Είναι κατακαιρματισμένη πολύ η εκπαίδευση. Το σύστημα βασίζεται κυρίως είναι, ε, ε, χρησιμοποιεί ακόμα πάρα πολύ χαρτί, δεν υπάρχει αρκετή ηλεκτρονική μηχανοργάνωση και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Επίσης, ε, είναι πολύ διαφορετικές οι αξιολογήσεις κινδύνου και οι πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι ε, το, τα κοινά ε, σύνορα που σε γενικές γραμμές θα πρέπει να προστατεύουν τον Ευρωπαίο πολίτη ε, πολλές φορές δίνουν πολλές δυνατότητες εκμετάλλευσης από τον κλάδο που γνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορές αντιμετώπισης από τα κράτη-μέλη. Όπως είπα και προηγουμένως, βασίζεται στα χαρτιά το σύστημα ε, είναι δύσκολο λοιπόν να παρακολουθήσει κανείς την έκδοση των πιστοποιητικών αλλιευμάτων και των δηλώσεων επεξεργασίας και όπως επίσης και το πόσο, κατά πόσο είναι αυθεντικά τα έγγραφα αυτά. Επομένως υπάρχουν περιπτώσεις διπλής χρήσης πιστοποιητικών. Ε, η μοίρα των φορτίων που απορρίπτονται δεν ε, είναι γνωστή, είναι διαφέρει ανάλογα με το κράτος μέλος. Ε, μερικά αποστέλλονται πίσω στη χώρα προέλευσης, μερικά χάνονται και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των κυρώσεων που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη και μια σημαντική, παραπολή, μια σημαντική πτυχή ενός τέτοιου κανονισμού είναι αποτρεπτικός χαρακτήρας του. Επομένως, αν οι κυρώσεις είναι διαφορετικές μεταξύ των κρατών μελών, ε, δεν παρουσιάζει συνοχή ο κανονισμός και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον έλεγχο των ε, επανεξαγωγών και επομένω υπανοσαγωγών ε, είναι ε, ανεπαρκής και εντελώς διαφορετικός από χώρα σε χώρα. Γιατί πολλέ φορέ κάτι, κάποιο φορτίο αποστέλλεται για επεξεργασία εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια πανισάγεται. Αυτό μπορεί να συμβεί δύο-τρει φορέ. Και αποτέλεσμα είναι ότι η ανιχνευσιμότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αυτή την περίπτωση και όλο και περισσότερο δυσχεραίνεται από αυτό το μη ηλεκτρονικό σύστημα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με ε, ε, φορτία σε τμήματα τα οποία πηγαίνουν σε διάφορες χώρες και μετά επιστρέφουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα τις εκθέσεις για τις δραστηριότητες ε, της Ένωσης ε, ε, των κρατών μελών και των πορισμάτων τρίτων χωρών, δεν είναι δημόσια γνωστές οι εκθέσεις αυτές κάτι το οποίο διευκολύνει την παρακολούθηση της εφαρμογή του κανονισμού και δεν μπορούμε να ξέρουμε και πόσο επιτυχής είναι. Είναι, σαφ, είναι κατά πόσο οι έλεγχοι γίνονται στις τρίτε χώρες και αν γίνονται οι έλεγχοι, ε, αν αντιμετωπίζουν, ε, αν όντως καλύπτουν ε, τα μέτρα ε, της σημαία, ε, του παράκτιου κράτους και τον ελέγχων που γίνονται από ε, τους λιμένες ε, στην αγορά κλπ. Η ανιχνευσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για την αποτελεσματική ε, εφαρμογή του κανονισμού και του προγράμματος πιστοποιητικών αλλιευμάτων, κάτι το οποίο, που το οποίο τίθεται να αμφιβόλα από τις διαφορές ελέγχων στις τρίτες χώρες από τη στιγμή της εκφόρτωσης μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής. Πρέπει να υπάρχει μια συνοχή στον έλεγχο. Ε, τα εθνικά ε, προγράμματα αντιμετώπισης της παράνομης αλληλείας, ε, μέτρα του λιμένα, των κρατών σημαίας, είναι εντελώς, διαφορετικές, είναι εντελώς διαφορετικός ο έλεγχος που γίνεται ανάλογα με τη χώρα για την οποία μιλάμε. Πολλέ ε, χώρες έχουν προβεί σε μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος ανιχνευσιμότητας, άλλε όχι. Οπότε υπάρχει μεν ε, μία ε, τάση βελτίωσης που έγινε στο πλαίσιο του κανονισμού για την παράνομη αλληλεία, όμως δεν είναι συνεπής η εφαρμογή του και σε πολλές περιπτώσεις τα μέτρα των κρατών μελών δεν είναι επαρκή για να ε, επιτευχθεί η, α, η ανιχνευσιμότητα. Η διαμετακόμιση τώρα δεν γίνονται έλεγχοι σε κάθε περίπτωση και γίνονται, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ε, για τη διαμετακόμιση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει σύγχυση, έλλειψη σαφήνειας ε, για το ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές, για την επικύρωση των πιστοποιητικών, ε, της μεταφόρτωσης στη θάλασσα ή ε, στο λιμένα, για τις δηλώσεις επεξεργασίας. Υπάρχει λοιπόν σύγχυση στον τομέα αυτό και δεν υπάρχουν και αντικειμενικά κριτήρια ε, για την, τον ορισμό του ποια αρχή είναι η αρμόδια για τις ε, συγκεκριμένες αυτές λειτουργίες. Ε. Και υπάρχουν έτσι και έμεσες εισαγωγές μη μεταποιημένων προϊόντων που μπορούν να εισαχθούν στη χώρα μέσω πιστοποιητικών τρίτων χωρών, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία αποδεικτικά ε, ελέγχων ε, παράκτιων ε, ή του κράτους λιμένα. Κάτι το οποίο βέβαια δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην παρακολούθηση και στην εποπτεία βάσει της διεθνούς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας. Σε μερικές περιπτώσεις τα τμήματα των φορτίων δεν ελέγχονται σωστά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση ε, της φόρμας ε, T2M που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα σκάφη για την εισαγωγή ε, των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φόρτωση και εκφόρτωση των αλλιευμάτων τους σε εμπορευματοκιβώτια σε τρίτες χώρες, γιατί τα T2M φορτία δεν υπόκεινται σε ελέγχους όταν πρόκειται για χώρες από τις οποίες έγινε η αλίευση ή όταν είναι χώρες διαμετακόμισης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν, ε, κάποια αλλιεύματα της ανοιχτής θάλασσας, για παράδειγμα, δεν υπόκεινται ε, σε χρήση πιστοποιητικού αλλιεύματος ή δήλωσης επεξεργασίας. Ε, αυτό είναι λόγω του κανόνα της προέλευσης, θα τον γνωρίζετε, ή του, είναι, είναι τελωνιακό θέμα. Ε, και την έλλειψη εφαρμογής ε, του γράμματος του, ε, κανονισμού για την παράνομη αλία. Ο ορισμός της εξαγωγής, για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου δεν συνάδει με αυτό που προβλέπεται στον κανονισμό για την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, η μελέτη μας παρουσιάζει 11 συστάσεις σε σχέση με την ε, υγειονομική συμμόρφωση και 23 συστάσεις ε, σε σχέση με την συμμόρφωση ε, με τον κανονισμό παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πέλιν. Δεν ξέρω αν η κυρία θέλει να παρέμβει ή όχι, η κυρία Γκοντά. Παρακαλώ, θέλετε να παρέμβετε κυρία Γκοντά. Όχι. Εντάξει. Ωραία, τέλεια. Θα κάνουμε ένα γύρο παρεμβάσεων τώρα. Η κυρία Φράγκα πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Πέλιν. Εγώ πρέπει να πω πρόεδρε ότι διαβάζοντας με προσοχή την έκθεση του πρέπει να πω ότι με εξέπληξε πολύ αρνητικά. Αυτό το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά, την ισπανική περίπτωση δηλαδή, τι συμβαίνει με την Ισπανία. Και τόσο πολύ εξεπλάγει που παρόλε τι προσπάθειε που έγιναν από την Ισπανία και που έχουν αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλου, και μια και αυτό το θέμα με ενδιαφέρει άμεσα και το γνωρίζω σε βάθο, διαπίστωσα πάρα πολλά σφάλματα, πάρα πολλά λάθη όσον αφορά την Ισπανία, τη χώρα μου. Και δεν ξέρω τι συμβαίνει για τι άλλε χώρε, αν έγινε αυτό η περιγραφή με τον ίδιο βαθμό σφαλμάτων και που βρίθουν εδώ. Πρώτα, αναλύοντας την ε, μεθοδολογία, ήθιστε σε τέτοιου είδους μελέτες που γίνονται σε επαφή με τα κράτη-μέλη, πάτε εκεί, συλλέγετε πληροφορίες, συζητείτε, και λόγω ευγένεια κιόλα και για να μπορεί να έχει κανείς και να ολοκληρώνει κάποια κενά που μπορεί να υπάρχουν στις εκθέσεις. Αυτό που γίνεται κανονικά είναι αποστέλλεται κανονικά αυτές τις εκθέσεις στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη κάνουν παρατηρήσεις που εσείς μπορείτε να λάβετε ή όχι υπόψη σας. Όμως, πραγματικά, εγώ ζήτησα από την Ισπανία να δω τι γίνεται και πληροφορήθηκα <clears throat> ότι πήραν την έκθεση όπως την πήρα και εγώ. Δηλαδή δεν μπόρεσαν να κάνουν σχόλια οι παρατηρήσεις, οι ισπανικές αρχές, ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί το κείμενο αυτό. Για αυτούς, για τους λόγους μπορώ να πω ότι δεν αντανακλάται η ίδια η πραγματικότητα της Ισπανίας, για παράδειγμα με την παράνομη λαθρέα λία. Σας ε, δόθηκαν τα στοιχεία τα οποία χρειάστηκαν, ε, ε, εφιστώντας την προσοχή στη δομή των ελέγχων, του τι γίνεται με τα τελωνία σε σχέση με τις υπηρεσίες εποπτείας αλίας, το μόνο που κάνατε εσείς και λέτε είναι ότι κάνετε λόγο για μια κεντρική διαμόρφωση διαχείρισης. Τίποτα άλλο δεν κάνατε. Για παράδειγμα, όσον αφορά την, τους επόπτες, την εποπτεία, εσείς λέτε ότι οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις γίνονται κατά τη διάρκεια ε, των Σαββατοκύριακων δεν γίνονται έλεγχοι. Πρέπει να σας πω ότι 365 μέρες το χρόνο γίνονται οι έλεγχοι αυτοί στην Ισπανία και οι ελεγκτές έχουν βάρδιες 15 ωρών δραστηριότητας. Πράγμα το οποίο στην έκθεσή σας φαίνεται ότι μια και το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι είναι όλοι ε, σε αργία και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό αντανακλάται στην έκθεσή σας. Λέτε ότι σε σχέση με την Ιβυρική Χερσόνησο ε, όσον αφορά συγκεκριμένους κανόνες για τα σκάφη καταλήγεται σε ένα συμπέρασμα που δεν συμμερίζομαι εγώ. Λέτε ότι είναι ένα παράδειγμα λέτε αυτό που δείχνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερο ζήλο και να κάνουν περισσότερους ελέγχους για τους τόλους τους. Αυτό δεν είναι παράδειγμα, δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο. Στην Ισπανία υπάρχει μόνιμη, ε, μόνιμη μέρημνα για τα σκάφη μας σε σχέση με τα αλλιεύματα, σε σχέση με την ε, ζώνη της Σιβηρίας και σε σχέση με άδεια αλλιείας που μπορεί να είχε εκδοθεί από μια ε, εταιρεία που μπορεί να υπέπεσε σε κάποια ολιστήματα ή απάτες. Τώρα, σε σχέση με τη Λιβερία που ε, αυτά τα θέματα ε, μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ Λιβερίας και ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κατανοώ πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υφίστανται αυτές οι παρατηρήσεις. Και όταν κάνετε λόγο για τους ελέγχους και διαπιστώσεις των πιστοποιητικών επανεξαγωγής, Εκεί όπου λέτε ότι η Γενική Γραμματεία Ελέγχου και ε, Επιθεωρήσεων με έδρα στην Μαδρίτη δεν έχει πλήρη στοιχεία σε σχέση με την, ε, τα ζητούμενα αυτής της έκθεσης στους λιμένες εισαγωγής. Και αυτό έχει επιπτώσεις ε, σε άτομα. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η μονάδα και για να ενημερωθούν όλοι έχουν, έχει πρόσβαση πέρα από τα πιστοποιητικά αλλιευμάτων και ε, δηλώσεις ε, μεταποίησης και σε υγειονομικά στοιχεία, στοιχεία μεταφοράς, ε, λογαριασμούς και πιστοποιητικά όπως χρειάζονται. Όλα αυτά για να πω ότι εσείς απλουστεύσατε υπερβολικά το έργο σας με τρόπο ανεπίτρεπτο. Σε άλλη σελίδα λέτε ότι σε σχέση με το ότι αναλύονται μόνο κάποια πιστοποιητικά ε, σύλληψης ε, αλλιευμάτων πρέπει εδώ να σας πω και να αναφερθώ αν θέλετε να το πάρετε ως αποδεικτικό στοιχείο μπορείτε να πάτε στην Ισπανία να δείτε δεν αληθεύει σε σχέση με τα αντίγραφα ε, και τα πιστοποιητικά τα οποία δεν υφίστανται υπάρχουν δηλώσεις τελωνίων και ίδια η άδεια αλληλείας που εκδίδεται. Αν είναι αναγκαίο να δει κανείς αν έχουν ε, υπερβεί τα, τις ποσοστώσεις ε, σε σχέση για παράδειγμα με τη σημαία του σκάφους, αυτά είναι θεμελιώδους σημασίας. Αυτά είναι κάποιες παρατηρήσεις που δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο ε, κανόνα λόγο για την περιβόητη έκθεση της ΝΟΑ, όπου για παράδειγμα λέτε εσείς ότι η Ισπανία λέτε αντιμετωπίζεται ως ε, ένα κράτος, ε, έχει μια στάση ως ένα κράτος το οποίο δεν είναι υπεύθυνο, δεν αληθεύει αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι βλέπω με άλλα λόγια στην ανάλυση σας υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα χάσματα και κενά μεθοδολογίας και αποτελεσματικότητας και ε, απόδοσης της αλήθειας. Σε σχέση με την παράνομη αλληλεία που υπάρχουν ίσως ε, ανάγκες να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες, δεν το αρνούμε αυτό. Σε σχέση όμως με το τι γίνεται για τα σκάφη ενός ε, κράτους μέλους όπως είναι η Ισπανία, αμφιβάλλω για την αληθεία και την πιστοποίηση αυτών των στοιχείων που αναφέρετε εσείς. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κυρία Λοβέν, παρακαλώ. Ε, thank ε, Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την μελέτη αυτή που δεν μπόρεσα ακόμα να τη διαβάσω, αλλά σίγουρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί εγώ ήμουνα η συγγήτρια για το πώς, στο θέμα πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιμετωπίσει την αλία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρότι λοιπόν μπορώ κάλλιστα να φανταστώ ότι και προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ε, του κανονισμού περί παράνομης και αναρχής ε, αλίας όταν πρόκειται για την ανιχνευσιμότητα. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι πρόκειται για ένα κομμάτι νομοθεσίας όπου αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην παγκόσμια λία, αρχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια κατάσταση, άρα δηλαδή ε, βρισκόμαστε ακόμα στα σπάργανα όσον αφορά τις επιπτώσεις ε, της ε, αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε άλλες αγορές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι και άλλοι παγκόσμιοι παίκτες να εφαρμόσουν παρεμφερή νομοθεσία η οποία θα καθιστά δυνατόν ε, τα, λαθρέα αλία και τα λαθρέα ψάρια να εμφανίζονται σε άλλες αγορές εφόσον δεν θα εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρετίζω βέβαια τις συστάσεις για βελτίωση πάνω σε όλα αυτά, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να ε, είναι κανείς υπερήφανος ε, για την ε, ευρωπαϊκή, την ενωσιακή αλία, πραγματικά αρχίζουμε να μετακινούμε διάφορα πράγματα σε τρίτες χώρες. Και διαβάζοντας την ομοθεσία για την παράνομη και άναρχια αλία, βεβαίως και πρέπει να συμφωνήσω ότι τα κράτη-μέλη καλούνται να ε, συμφωνήσουν ε, στις καλύτερες επιδόσεις και ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ενδεχομένως ε, να εμφανίζονται στον κατάλογο της παράνομης λατρείας και ανερχής ε, αλίας. Ίσως πράγματι πρέπει κάνα να ε, καταργήσουμε κάποια ε, επιδόματα που χορηγούνται γιατί ίσως με τον τρόπο αυτό να περιοριστεί και η παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδράσεις ε, για τις συστάσεις που έχουν προκύψει από αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Στρομέβα, παρακαλώ. ευχαριστώ πρέπει να πω δεν μπόρεσα να μελετήσω αυτή την έκθεση ακόμα. Παρακολουθούσα αυτά τα θέματα και ωστόσο για κάποια ερωτήματα, κάποια σχόλια τα οποία πρέπει ε, να γίνουν όσον αφορά την ε, ουσία αυτή. Γενικά Έχω κάποιες αμφιβολίες πρέπει να πω, κάποια ερωτηματικά που θα ήθελα να θέσω, ε, κάποια ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα για το τρέχον σύστημα και ουσιαστικά για το ρόλο της, ε, ε, του τι γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ για τον καθορισμό κανόνων και διατάξεων ώστε τουλάχιστον να μπορούν να γίνονται δεκτά τα όσα υποβάλλονται από τις υπόλοιπες χώρες ως στοιχεία, ενώ έχουμε διάφορες περιπτώσεις όπου τα όσα διατίθενται από κράτη-μέλη συμπεριλαμβάνουν πολλές φορές ακόμα και εκείνα τα οποία δεν υλοποιούν τις βασικές αρχές που θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες όσον αφορά τις προϋποθέσεις ε, για την υγιεινή και τις ε, διατάξεις για την εργασία. Συγκεκριμένες χώρες που μπορούμε να ε, αναφέρουμε, Κίνα και άλλες, το πρόβλημα είναι ότι εκεί το σημερινό σύστημα δεν μας επιτρέπει να κάνουμε ελέγχους, να επιθεωρούμε, να εποπτεύουμε, δεν μας επιτρέπει να, μας επιτρέπει να αντιδράσουμε και να δράσουμε. Και έτσι το θεωρούμε ως δεδομένο και το δεχόμαστε αυτό με έναν τρόπο που δεν μπορεί η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ να κάνει τίποτα άλλο παρά για παράδειγμα να προσπαθήσει να βρει κάποιες ίσως εναλλακτικέ δυνατότητες για να σταματήσουν ε, κάποιες δραστηριότητες σε σχέση με αυτά τα σκάφη. Έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα και από άλλες εκθέσεις ε, και βλέπουμε ποια είναι η εμβέλεια αυτού του, του προβλήματος. Παρόλα αυτά η, ΣΑΝΚΟ δεν είναι σε θέση να αντιδράσει όπως πρέπει. Ερώτηση λοιπόν, ερώτημα. Επειδή α, καθώς είδα το κεφάλαιο για, που αφορά την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, ίσως ε, αυτό το θέμα ε, δεν αναφέρει το όπως θα έπρεπε και ιδιαίτερα όσον αφορά τον κανονισμό για την καταπολέμηση της ε, ε, λαθρέας αλίας, παράνομης αλίας. Ε, συμφωνώ με την παρατήρηση αλλά και για τη γενικότερη αντίληψη ότι πρόκειται για ένα κέριο μέσο και εργαλείο που είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε οπωσδήποτε στις διάφορες δράσεις μας ε, για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, όχι μόνο ένα ερώτημα για το πώς θα υλοποιήσουμε όλα αυτά τα μέτρα, πράγμα που είναι σημαντικό αυτού αλλά και το θέμα των επιπτώσεων όλων που συνεπάγονται αυτά για το σύστημα αυτό και την εφαρμογή του και τις επιπτώσεις που έχει σε άλλες χώρες. Λαμβάνομαι υπόψη για παράδειγμα ότι έχουμε την υποχρεωτική ας πούμε συμμόρφωση των βιομηχανιών και των επιχειρηματιών με τους κανονισμούς και κανόνες αυτούς. Τώρα όλα αυτά προκαλούν και κάποιες αλλαγές τουλάχιστον στο νομικό πλαίσιο αυτών των χωρών που λαμβάνονται υπόψη. Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα υπάρχει, υπάρχουν επιπτώσεις και σε μεγάλο βαθμό δεν είναι τέλεια όλα αυτά, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να σημειώσουμε για τις συστάσεις για παράδειγμα, βλέποντάς τις, προσπαθώντας να δούμε αν αυτή η προοπτική μπορεί έτσι να ληφθεί υπόψη ή όχι, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωση, την ιδέα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Η ιδέα ουσιαστικά είναι ότι δεν έχουμε τα μέσα, τα εργαλεία, δεν έχουμε το πραγματικό δυναμικό για να υπάρξει η συμμόρφωση από πλευρά των άλλων, των τρίτων. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν μέσων εργαλείων, κονδυλίων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και διαφορετική προσέγγιση αυτών των προδιαγραφών σε σχέση με άλλες χώρες που είναι που ε, υφίστανται τις επιπτώσεις ε, των αλλιευμάτων αυτών αλλά και εκείνων που εμπλέκονται περισσότερο σε σχέση με τη συνιστόσα των αγορών. Έτσι λοιπόν μπορεί αυτή η ομάδα χωρών να αποτελέσει ε, αντικείμενο να μπορέσουμε τη συζήτηση αυτή να την εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτό το γενικό πλαίσιο. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που ήθελα αρχικά να θέσω. Ίσως μπορεί να υπάρχουν κάποια από αυτά τα στοιχεία στην έκθεση, αλλά δεν τα εντόπισα εγώ. Και αν μπορείτε αυτά να μας τα διευκρινίσετε, αυτά που ανέφερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Ντέιβις, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ και για την έκθεση αυτή γιατί ε, είναι ένας πολύ ωραίος κατάλογος για το τι πρέπει να κάνουμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Ε, καταρχήν, όσον αφορά τα σχόλια της κυρίας Φράγκα όπου επισημαίνει διάφορες ασάφειες ε, εγώ τα διάβασα όλα αυτά και δεν είμαι σίγουρος αν λειτουργεί το σύστημα. Δεν έχω αυτές τις ε, γνώσεις. Εσείς είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με κάποιους ε, που υποτίθεται ότι εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες κυρίως με την Κομισιόν. Λένε αυτή είναι η σύσταση που κάνουμε. Αλλά εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι να εντοπίσει κανείς τις αδυναμίες στη σύσταση και ορισμένα αυτά τα πράγματα, παρότι έχουν πάρα πολύ ωραία, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι στην πρακτική πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Εύκολο, εύκολα λέγεται ότι πρέπει να γίνει κάτι, αλλά μερικές φορές δεν είναι εύκολο να γνωρίζει κανείς πώς μπορούν να γίνουν στην πράξη όλα αυτά. Και διερωτώ με σχετικά με τη χρηματοδότηση όσον αφορά αυτή τη σύσταση ε, για την αλία, ε, την παράνομη, τη και την άναρχη. Ε, να σταματήσει η χρηματοδότησή της, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτά σχετίζονται και με τη συζήτηση που επίκειται σχετικά με το, τις μηχανές, το μέγεθος των μηχανών και ούτω καθεξής. Και τέλος, όσον αφορά τον φορέα ελέγχου της αλίας. Δεν ξέρω, έχετε μιλήσει μαζί τους, ε, σας είπαν ε, τη γνώμη τους για όλα αυτά τα θέματα. Μήπως υπάρχουν ε, κάποιοι περιορισμοί ε, δεν βλέπω να υπάρχουν ε, συστάσεις σχετικά με το ρόλο αυτού του φορέα στην αντιμετώπιση της ε, παράνομης λαθρέας και αναρχής ενέργειας. Σας ευχαριστούμε. Έγινε ο πρώτος γύρος. Θα λάβει τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε σε αυτή τη συνεδρία να συμμετάσχουμε. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβάσαμε με πολύ ενδιαφέρον αυτή την έκθεση και επίσης σίγουρα προσέξαμε τις παρατηρήσεις του εισηγητή στην παρουσίαση που έκανε απόψε. Γνωρίζουμε και αυτό είναι η αφετηρία μας ότι ο κανονισμός κατά της λαθρέας και παράνομης αλληλείας παρόλες τις προόδους που σημειώνονται δεν είναι ένας τέλειος κανονισμός σε σχέση με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για κάθε έναν με τις ευθύνες που πρέπει να επομίζεται, δεν είναι τέλειο το πλαίσιο. Το γνωρίζουμε αυτό. Πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα. Με αυτοκριτική αντιμετωπίζουμε τα πράγματα έναντι των δράσεών μας. Αυτό είναι ένα γεγονός. Υπάρχουν πράγματα που σίγουρα μπορούν να βελτιωθούν σε αυτόν τον κανονισμό. Εντάξει, σίγουρα. Άλλο πράγμα τώρα είναι ότι πολλές από τι επικρίσεις που διατυπώνονται σε αυτή την έκθεση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα κράτη-μέλη για αυτόν τον κανονισμό, ότι αληθεύουν όλες οι επικρίσεις. Όχι, δεν συμφωνούμε. Έχουμε και εμείς ε, κριτική τοποθέτηση όσον αφορά με αρκετό μέρος της μεθοδολογίας. Αν θέλετε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, να επισέλθουμε Πρόεδρε. Αλλά θα ήθελα μόνο κάποια παραδείγματα να αναφέρω. Θεωρούμε ότι ένα τμήμα της μεθοδολογίας και ανάλυσης μόνο που κάνουν οι σύμβουλοι δεν αναπτύσσεται με καλό τρόπο και δεν έχει αναπτυχθεί καλά. Είναι το τμήμα που αφορά τους τελωνιακούς ελέγχους. Αυτό το τμήμα ε, αν επαρκώς έχει ε, διατυπωθεί και αναπτυχθεί και μια σειρά ανακριβιών αναφέρονται που δυστυχώς μας κάνει να αμφισβητήσουμε κάποια και από τα συμπεράσματα της ίδιας της έκθεσης. Μετά στη συνέχεια υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία θεωρούμε ότι χρειάζονται διευκρινήσεις. Παράδειγμα, λέγεται ότι παράδειγμα, ότι δεν γνωρίζουν λέει πολύ καλά αν η έλεγχη που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναφερθεί μια χώρα ως χώρα παράνομης και λαθρέας αλίας είναι αλλίας Και εδώ έχουμε το αίτημα που ε, δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει οκτώ χώρες ως μη συνεργαζόμενες χώρες ε, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης λαθρέας αλλίας. Εδώ υπάρχουν διάφορα θέματα από πλευρά σκεπτικών και θεωρούμε ανάλυση η οποία είναι ευρύτερη. Γιατί λοιπόν είτε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι πλήρη η έλεγχη ή όχι. Πρέπει με βάση τα όσα έγιναν να μα πούν τι είναι εκείνο το οποίο ε, απουσιάζει η λύπη. Επίσης λέγουν ότι πιστοποιείται ότι στους φακέλους που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει αδιαφάνεια, θολός ε, χαρακτήρας ε, ε, στα, στα στοιχεία που εξετάζονται. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Είμαι φυσικά πρόθυμος για άλλη μια φορά να εξηγήσω όλα αυτά γιατί η ροή των πληροφοριών φυσικά πρέπει να είναι περιορισμένη υπό εχεμήθεια ή υπό διατήρηση του απορρίτου για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα υπεράσπισης ε, νομικά και δικαστικά των ε, όσων κατηγορούνται. Γι' αυτό πολλές από τις πληροφορίες ε, που υπάρχουν για να δημιουργηθεί, να τεκμηριωθεί μια περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι άλλου κράτους, πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα στοιχεία ως εμπιστευτικά στοιχεία που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Γιατί αν δημοσιοποιούνται τότε θα έχανε την αποτελεσματικότητά της η προσφυγή αυτή. Δεν είναι λοιπόν καμιά βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι θολή η διαφανής είναι απαραίτητο στοιχείο και αναγκαίο στοιχείο η εχεμήθεια και το απόρριτο για να μπορέσουν αυτά τα στοιχεία να ευδοκιμήσουν στο τέλος. Λέτε μετά ότι οι επιδοτήσεις ε, μπορούν να αυξήσουν λέει, την εμβέλεια της ε, παράνομης και λαθρέας αλίας. Δεν υπάρχουν ε, λοιπόν και ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιες επιδοτήσεις. Πρέπει εδώ να αποσαφηνίσουμε ότι στην Ολομέλεια στις 22 Οκτωβρίου θα συζητήσετε μια έκθεση για τις επιδοτήσεις, ενισχύσεις για την αλία και φαντάζομαι ότι δεν είναι όλες, δεν θα είναι όλες οι ενισχύσεις και επιδοτήσεις κάτι αρνητικό. Δεν μπορεί λοιπόν να πει κανείς ε, ότι κάτι τέτοιο ε, ισχύει ισοπεδωτικά. Ή θα πρέπει λοιπόν να διαφοροποιήσουμε ή δεν θα αληθεύουν όλα αυτά. Είναι κάποια λίγα παραδείγματα πρόεδρε που δείχνουν ότι έχει κάποια θετικά και ενδιαφέροντα στοιχεία η έκθεση. Για παράδειγμα γίνεται ε, διατυπώνεται η παρατήρηση ότι ένα σύστημα που βασίζεται στην έγγραφη, έντυπη μορφή ε, ευνοεί τις απάτες ε, και τα ολιστήματα. Σε αυτή την περίπτωση συμφωνούμε, εντάξει. Κάνει μια σωστή ανάλυση η μελέτη ότι όλα τα συστήματα τα οποία ε, θεμελιώνονται σε έντυπη ή έγγραφη μορφή, εντάξει, έχουν αυτά τα λατώματα. Όμως ε, οι διοικήσεις, οι αρχές των κρατών μελών μας είπαν για να πάμε σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, πράγμα το οποίο όλοι επιθυμούμε, χρειάζεται χρόνος και χρειάζονται πολλά κονδύλια. Και αυτό θα είναι μια μεταγενέστερη φάση στην ανάπτυξη των ε, πρωτοβουλειών μας. Ε, και αν ε, είναι κάτι για το οποίο συμφωνούμε στην ανάλυση μπορεί να είναι αυτό. Δεν ξέρω τώρα Πρόεδρε να υπησέλθουμε σε μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομεριών, πιο εξειδικευμένα. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να το κάνουμε αν επιθυμείτε. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτής της μελέτης. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι εμείς υλοποιούμε μια μελέτη που θα είναι έτοιμη ιστερότερα κατά τη διάρκεια του έτους και πάλι θα δοθούν πρόσθετα στοιχεία πληροφοριών για εκείνες οι πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν. Είτε είναι για τον ίδιο τον κανονισμό αυτό, είτε για την πρακτική εφαρμογή διατάξεων και ε, συγκεκριμένων ρητρών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Είμαστε πρόθυμοι από την Επιτροπή να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με τον πιο παραγωγικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα. Ο κύριος Ρωμέβα, επειδή με ενέπνευσε ο συνάδελφος, ε, ίσως λοιπόν το ένα πρόβλημα είναι να πει κανείς ότι να το θέσουμε συζήτηση ότι ο κανονισμός καταπολέμησης της παράνομης λαθρέας ε, αλίας δεν είναι το θέμα να απαγορεύσουμε τις εισαγωγές, δεν είναι ο τελικός στόχος ενός τέτοιου κανονισμού, αλλά να αλλάξουμε την συμπεριφορά στην αλία των αλιέων την αλληλευτική συμπεριφορά. αυτό θα ήταν ο, ο μεγάλος μείζον η μεγάλη πρόκληση για να δούμε αν μια τέτοια ρύθμιση από πλευρά νομική είναι καλή ή όχι και θα μπορούσε να επεξηγήσει όλη αυτή την προσέγγιση που υιοθετούμε κάποιοι από εμά σε σχέση με αυτά τα θέματα. Αυτό για διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σύμφωνοι. Ευχαριστώ για αυτές τις επεξηγήσεις και για την έκθεση αυτή για την οποία υπάρχουν πολλές επικρίσεις. Έχετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Uh, perhaps um, address the comments or uh, Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, με τη σειρά με την οποία ετέθησαν. Ε, ως προς τη μεθοδολογία, κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να κάνουν τέτοιου είδους εκθέσεις, ε, η μεθοδολογία συμφωνήθηκε με την γραμματεία της Επιτροπής σας και Υποθέτω ότι ακολούθησε τη συνήθη μεθοδολογία που συνήθως ε, ακολουθεί η Επιτροπή, ε, η σας. Ε, δεν είχε αναφερθεί ποτέ ότι έπρεπε να λάβουν τις εκθέσεις αυτές τα κράτη-μέλη. Εμείς αυτό είχαμε συμφωνήσει με τη Γραμματεία και αυτό εφαρμόσαμε. Τώρα κατά πόσο θα, θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να τα λαμβάνουν τα στοιχεία αυτά ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση του σκάφους ε, στη Λιβερία, αυτό είναι κάτι ε, το οποίο υπάρχει στα, στη βιβλιογραφία μας ε, και υπάρχουν και οι σχετικές πηγές. Τα κράτη-μέλη υποκύπτουν μερικές φορές τον πειρασμό της παράνομης, λαθρέας και άναρχης αλίας και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τις δραστηριότητες ε, στόλων που αλλιεύουν ε, πολύ μακριά, σε μακρινές αποστάσεις γιατί υπάρχουν τα μέτρα του ε, κράτους ε, ε, σημαίας, αλλά μερικές φορές παρεκκλίνουν των μέτρων του κράτους λιμένα ε, ή του παράκτιου κράτους. Οπότε γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί Υπάρχουν διεθνείς προδιαγραφές ε, παρακολούθησης, υπάρχουν μέτρα λιμένα, κράτους σημαίας, παράκτιου κράτους ε, και αγοράς. Αυτή, αυτή, αυτά τα τέσσερα είδη μέτρων υπάρχουν και σας παρατρύνω όλους να είστε προσεκτικοί επί των ε, σημείων αυτών. Δεν αρκούν μόνο τα μέτρα του κράτους σημαίας. Όσον αφορά τώρα την ε, διαχείριση του προγράμματος ε, πιστοποιητικών αλλιευμάτων, είναι κεντρικό το σύστημα από την περιφέρεια της χώρας από διάφορους λιμένες ε, εισάγονται τα προϊόντα και είναι γεγονός ότι λαμβάνουν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα και ενδεχομένως ε, αντίτυπα του μεγαλύτερου τμήματος του πακέτου. Αλλά η τεχνική ε, μου άποψη είναι ότι οι έλεγχοι γίνονται καλύτερα στο λιμένα εισόδου. Γιατί εκεί μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει το σύνολο των εγγράφων που είναι διαθέσιμα τη στιγμή της εισόδου, στο σημείο της εισόδου ε, και επίσης μπορεί κανείς να κάνει και ε, ελέγχους επιτόπου όταν, αισθάν, όταν νιώθει κάτι δεν πάει καλά. Ε, αυτή είναι η δική μας τεχνική άποψη. Ενδεχομένως η Ισπανία να είναι ικανοποιημένη με τις ε, επιδόσεις της, αλλά πιστεύουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ε, έχει βελτιωθεί και μερικά κρατημέλη τα έχουν καταφέρει. Όλα αυτά είναι όμως απλώς παραδείγματα του πόσο ε, σας οικετεύουμε να είστε προσεκτικοί για τα θέματα αυτά. Μην, μην εφησυχάζετε. Δεν υπάρχει ποτέ τέλειος έλεγχος, δεν τα ελέγχετε όλα και πάντοτε υπάρχει περιθώριο ε, βελτίωσης. Υπάρχει και κάτι άλλο που αφορά τα κράτη-μέλη. Εμείς δεν κάναμε πλήρη έρευνα και δεν μας ζητήθηκε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να τον, απλώς τονίσαμε ζητήματα που πιστεύουμε ότι πρέπει να εξεταστούν. Και ένα από τα ζητήματα που τονίσαμε δεν ήταν η έλλειψη εναρμόνισης των πρακτικών, ε, αλλά το γεγονός ε, ότι κάποια κράτη μπορεί να συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο από κάποια άλλα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι κατά πόσο συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη χώρα ή αν είναι η γραμματεία της συγκεκριμένης χώρας. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επί των σημείων αυτών. Να Εντοπίζουμε την απάτη, τις ύποπτες δραστηριότητες ε, και να εξασφαλίζουμε βέβαια την τήρηση των κοινών συνόρων χωρίς βέβαια να ε, πλήττουμε την αυτονομία των κρατών μελών. Δεν προσπαθούμε λοιπόν να δείξουμε με το δάχτυλο συγκεκριμένες χώρες, απλώς δίνουμε παραδείγματα που πιστεύουμε ότι δείχνουν ακριβώς αυτές τις ανησυχίες που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας άναρχης Κυρία Λεύιν... Αναγνωρίζω ότι είναι ένας ε, μοναδικός ε, κανονισμός, είναι καινούριος, δεν το τόνισα ενδεχομένως ε, στην έκθεση επαρκώς, αλλά το είπα στην αρχή της παρουσίασής μου, ότι το υγειονομικό κανονισμός είχε κάποιο χρόνο να οριμάσει, ενώ ο κανονισμός για την παράνομη αλία είναι καινούριος εντάξει, το αναγνωρίζω. Ε, είχαμε πολλά πράγματα να εξετάσουμε σε σχέση με τον κανονισμό της παράνομης αλίας. Δεν θέλουμε να διατυπώσουμε. Θέλουμε απλώς να κρούσουμε κόδωνε κινδύνου και να εντοπίσουμε προβλήματα για την ε, διαδικασία εφαρμογής που ο κύριος Πένια με μεγάλη ειλικρίνεια ε, ανέφερε. Ε, ήταν ειλικρινής ε, ως προς το ότι υπήρξαν, ε, υπάρχουν αδυναμίες στον κανονισμό για την καινούριο και μπορεί να βελτιωθούν οι διαδικασίες, αλλά μόνο αν ειλικρινώς αντιμετωπίσουμε, εντοπίσουμε κάποια προβλήματα που όντως υπάρχουν και τα αναγνωρίσουμε ως τέτοια. Όσον αφορά τώρα το θέμα της διαφάνειας, Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες πληροφορίες στο κλάδο που μπορούν ε, τέλος πάντων να ε, μαγειρεύονται με κάποιο τρόπο στο ένα ή στο άλλο δικαστήριο. Καταλαβαίνω ότι μερικές φορές υπάρχουν κάποια ζητήματα με τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ή άλλες γενικές διευθύνσεις σε σχέση με τον εφαρμογή του κανονισμού. Όμως πιστεύω ότι η οι πληροφορίες οι οποίες λάβαμε ε, μας δέδυναν τη δυνατότητα να ε, καλύψουμε το κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά ο κανονισμός ε, και μέχρι τις 29 Οκτωβρίου βάσει άρθρου του κανονισμού θα υπάρξει και σχετική έκθεση αξιολόγηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλοι φορείς της Επιτροπής θεωρούν ότι πρέπει να δημοσιεύονται εκθέσεις ελέγχου για 8 χώρες για παράδειγμα που αναφέρονται στον κατάλογο θεωρούν ότι πρέπει να αναφερθούν αλλά για άλλε επισκέψει σε άλλες χώρες ε, όπου οι ε, αρμόδιες αρχές ε, δέχτηκαν τις επισκέψει αυτές ή όχι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Υπάρχει μια ολόκληρη λοιπόν συζήτηση για την παράνομη αλία. Η ποιότητα Τη συζήτηση αυτή μπορεί να βελτιωθεί ίσως ε, εκδίδοντας λίγο περισσότερα στοιχεία, δημοσιεύοντας περισσότερα στοιχεία για το, για το θέμα αυτό που καλούμαστε να εξετάσουμε. Οπότε το λέω αυτό στο πνεύμα του να προχωράει κανείς ε, με μια ανοιχτή, σε μια ανοιχτή και ειλικρινή βάση. Δεν το λέω ούτε για να κατακρίνω. Είπα απλώ ότι είχαμε ένα πρόβλημα σε σχέση με τις πληροφορίες. Ε, πρέπει να έχουμε τις πληροφορίες για να μπορούμε να πούμε αντικειμενικά τι συμβαίνει. Α πούμε, ε, για τις, την απόρριψη ο κύριος Ρωμέβα με ρώτησε ποιος είναι ο αντίκτυπος της, του κανονισμού αυτού ε, ως τώρα. Μα δεν έχουμε τα σχετικά στοιχεία, δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία, δεν ξέρουμε. Οπότε μία από τις εκκλήσεις που κάνουμε είναι περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη τεκμηρίωση σε σχέση με το τι γίνεται. και νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορούν να ε, διατεθούν ως πληροφορίες ε, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα με οποιαδήποτε υπόθεση που είναι στο δικαστήριο οποιασδήποτε χώρας. Νομίζω ότι το κάλυψε αυτό το θέμα επαρκώς. Όσον αφορά τώρα το ρόλο της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, ΣΑΝΚΟ και τον κατάλογο των σκαφών, ναι, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τους ε, καταλόγους που, διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές. Πάντως τον FBO στέλνει αποστολές, πηγαίνουν στις εγκαταστάσεις, πηγαίνουν στα σκάφη, πηγαίνουν σε εγκαταστάσεις ε, επεξεργασίας, μεταποίησης. Τώρα το κατά πόσο το κάνουν αυτό αρκετά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δισταθμίσει κανείς βλέποντας ε, το όφελος, το κόστος ε, και το κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι μάλλον χαμηλός, οπότε από τεχνικής καθαρά απόψεως, δηλαδή μπορεί να θέλει κανείς μεγαλύτερη πειθαρχία από κάποιες αρχές, είπαμε ότι είναι λίγο ε, πρόχειρα τα πράγματα. Πρέπει το κράτος μέλος να αποφασίσει εάν επιπλέον, ε, ε, εάν, εάν επιπλέον, επιπλέον πόροι για να είναι μεγαλύτερη πειθαρχία πρέπει να διατεθούν ή όχι. Ενδεχομένως κάποιοι πόροι να χρειάζονται περισσότερο όχι στο υγειονομικό κομμάτι αλλά στο κομμάτι της παράνομης αλίας. Εκεί είναι που ε, χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους. Για τον αντίκτυπο λοιπόν που ρώτησε και ο κύριος Ρωμέβα δεν γνωρίζουμε και βεβαίως ε, ο κανονισμός δεν έχει σκοπό να σταματήσει τις εισαγωγές. Όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση και τη σχέση μεταξύ των επιδοτήσεων και της παράνομης αλληλείας, δεν νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες ε, ε, του τι σημαίνει αυτό από οικονομικής απόψης, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις που ενθαρρύνουν ε, υπερβολικές αλλιευτικές δραστηριότητες ε, μπορούμε βέβαια να το συζητήσουμε. Υπάρχουν πάντως ε, στοιχεία που υποστηρίζουν ε, την άποψη αυτή και είναι κάτι που γνωρίζω ότι ανησυχεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό επανεπισημαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η πτυχή, αλλά δεν είναι τεράστιο ζήτημα. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε να απάντησα στα ερωτήματα του πρώτου αυτού γύρου της συζήτησης. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, παρατήρηση κύριε Ρωμέβα. Δύο ουσιαστικά. Πρώτον, υπό τους όρους τακτικών ελέγχων ή επισκέψεων, η γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει ικανότητα για να γίνονται επισκέψεις ή επιθεωρήσεις στα σκάφη τα ίδια. Είναι σαφές αυτό. Και τα περισσότερα, οι περισσότεροι δεν πάνε ούτε καν στο λιμένα. Και εκεί υπάρχει μείζον πρόβλημα. Δεύτερον, Όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα εκεί. Δεν υπάρχει νομική ικανότητα για την τροποποίηση του πίνακα, να διαγραφούν, να βγουν κάποια σκάφη από αυτόν τον κατάλογο αν υπάρχουν υποψίες ή αν υπάρχουν και τεκμήρια και αποδείξεις ε, ότι δεν αλλιεύουν και δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις. Το μίσων, πρόβλημα δεν είναι η απουσία δυναμικού ελέγχων και ε, επιθεωρήσεων. Δεν υπάρχει και ούτε η δυνατότητα διοικητικά να βγουν κάποια πλοία από τους, ε, τον κατάλογο. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση έτσι σε αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Σημείο 9. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό έχει αποσυρθεί. Πάμε στα διάφορα. Στο 10 δεν υπάρχει κανένα θέμα ειδικό για τα διάφορα. Ανακοινώσεις του Προέδρου σε σχέση με τις αποφάσεις των συντονιστών. Εδώ υπήρχαν ένα ή δύο θέματα τα οποία εκκρεμούσαν καταρχήν. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με την Task Force όπως είχαμε πει. Καταρχήν διατηρείται, διατηρείται όπως είχαμε συμφωνήσει στη συνεδρίαση <clears throat> για τις 23 στις 4 το απόγευμα που θα είναι πρόεδρος, θα προεδρεύσει ο αντιπρόεδρος και τότε θα εξεταστούν ποια είναι τα θέματα για την Task Force, ποιο είναι το πρόγραμμα <clears throat> και με τον κύριο Πένα που ε, θα οδηγήσει αυτό το θέμα στην Επιτροπή πρέπει να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θα εργαστούμε, πώς θα δουλέψουμε σε σχέση με την επίσκεψη που θα κάνουμε, την αποστολή μας και θα δούμε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πιθανών συνεδριάσεων. Καταρχήν δεν υπάρχει άλλο θέμα σχετικά. Και με την έκθεση τώρα, τέλος, το σημείο 6.3 των συντονιστών σε σχέση με την έκθεση για την συμφωνία με την Κυριμπάτη, το κράτος Κυριμπάτη το έθετε η, Επιτροπή γιατί δεν, γνωρίζαμε σε σχέση με τη συνάντηση των συντονιστών αν υπήρχε δυνατότητα να ζητηθεί να συνταχθεί η σύνταξη έκθεσης από πλευράς των νομικών υπηρεσιών για το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτό το πρωτόκολλο. Και δεν είναι φυσικά απόφαση των συντονιστών και θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς με αυτή τη συμφωνία από πλευράς της ίδιας της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής. Και καταρχήν μου είπαν, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, ότι κυρία Λέβιν, εσείς έχετε τον λόγο να μας πείτε τα σχετικά, παρακαλώ. Ε, thank you, Chair. We had a very brief... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε μια σύντομη συνάντηση των σχεδόν πριν από την Επιτροπή. Δυστυχώς η συνάντηση αυτή ήταν πολύ μικρής διάρκειας και αυτό που αποφασίσαμε ήταν ότι οι σκιώδεις της συμφωνίας με την Κυριμπάτε θα συναντηθούν ε, τη μέθε επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν περισσότερο σε βάθος ε, το θέμα αυτό. Άρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό σήμερα στην Επιτροπή μας. Πολύ καλά λοιπόν. Από ό,τι καταλαβαίνω σε δύο εβδομάδες θα συνέρθετε, θα το δείτε αυτό υπό επιφύλαξη ότι όλα φυσικά ακολουθούν την κανονική τους διαδικασία σε σχέση με τα όσα μπορούν να εξελιχθούν μέσα σε δύο εβδομάδες. Θα πρέπει να το ξαναδεί λοιπόν η ίδια η Επιτροπή αυτό. Εντάξει, σωστό. The, shadows agreed to discuss it. Οι σκιώδες αποφάσισαν να το συζητήσουν ε, σε μια συνάντησή τους ε, σε δύο εβδομάδες τότε θα λάβουμε την απόφαση. Επειδή όμω υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί, η κυρία Πετρανίβη δεν θα είναι στι Βρυξέλλες, γι' αυτό ακριβώ θα πάρει τόσο χρόνο. Θέλουμε να το συζητήσουμε με όλους τους κοιόδους εισηγητέ Τέλεια, πολύ καλά. Λοιπόν, Εν πάση περιπτώσει θα την λάβει υπόψη να, η, θα λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή για το ποιο είναι αρμόδιο για την λήψη απόφαση. Εντάξει, σύμφωνοι. Κάποιο άλλο θέμα σε σχέση με αυτό το θέμα των συντονιστών δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση. Λοιπόν, παραμένουμε όπως συμφωνήσαμε. Η επόμενη συνεδρίαση 3 Οκτωβρίου, 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ, δεν υπάρχει άλλο θέμα. Λίγη συνεδρίαση, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και του διερμηνείς όπως πάντα. Γεια σας.